Αξιότιμοι συνάδελφοι, το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου πριν από 75 χρόνια ξεκίνησε ο δεύτερος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την επίθεση της Γερμανίας στη γειτονική χώρα της ναζιστικής Γερμανίας, στη γειτονική χώρα την Πολωνία. Ε, μια τραγική ιδεολογία με καταστροφικές τάσεις ε, ε, η τρέλα της ε, κατάκτησης ε, να επεκταθεί το Lebensraum σε γειτονικές χώρες. Άλλα κράτη έπρεπε να υποταχθούν, να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση, να υποδουλωθούν, ολόκληροι λαοί να εξαφανιστούν. Προέκυψε λοιπόν μια ακραία πολιτική που οδήγησε σε αυτό που αποκαλούμε ολοκληρωτικό πόλεμο είχε προηγηθεί ε, μια κοινική συμφωνία ανάμεσα στο Χίτλερ και το Στάλιν που οδήγησε ότι στην Πολωνία θα εισέλθουν και θα εισβάλλουν δύο στρατοί. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η Γερμανία εισέβαλε στη Ρωσία επέφερε τεράστια οντίνη στη χώρα αυτή με αποτέλεσμα μετά από έξι χρόνια το σύνολο της Γερμανίας δεν είναι πλήρως κατεστραμμένο. Μιλάμε για 60 εκατομμύρια νεκρούς. Πολλοί έπεσαν στο πεδίο της μάχης, ε, πέθαναν από την πείνα, ε, είχαν συλληφθεί, ε, άμαχος πληθυσμός, ηλικιωμένοι, παιδιά, γυναίκες, πολλοί που συστηματικά και με δόλο και σκοπό δολοφονήθηκαν, εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Πολλοί, όπως σας είπα, έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Είδαμε και την καταστροφή από βόμβες, από ε, ομοβροντίες. Πολλοί άνθρωποι εξάλλου ε, κρεμάστηκαν και πολλοί άλλοι έχασαν τη ζωή τους ε, στα, στους εξόντωση εξόντωσης ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα λοιπόν, μέχρι και σήμερα ζούμε υπό τις επίρειες αυτής της κατάστασης, αυτού του ρήγματος στον πολιτισμό. Θυμόμαστε όλες αυτές τις ε, φρικαλές πράξεις ε, και πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι 70 χρόνια μετά από αυτό το ρήγμα στον πολιτισμό επικράτησε η λύθη. Κάθε άλλο, σήμερα όλοι μας εξακολουθούμε να υποφέρουμε υπό τις επιπτώσεις αυτού του ολέτριου πολέμου και των προεκτάσεών του. Υπάρχει ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει από αυτόν τον πόλεμο. Ήταν η βούληση των γενεών που επέζησαν του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου να δημιουργήσουν δημιουργήσουν μια τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη που θα εμποδίζει επανάληψη τέτοιων πολέμων. Μιλάμε για την ε, διασυνοριακή συνεργασία πέρα από τα σύνορα, πέρα από οικονομικά, φυσικά, πολιτισμικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά σύνορα. Η βούληση λοιπόν να υπάρξει αυτή η συνεργασία, αυτή είναι η βούληση που ε, σφυριλάτησε την Ευρώπη που βιώνουμε σήμερα. Είναι η βούληση αυτή που οδήγησε και στην ε, κοινοβουλευτική μας συνέλευση. Εδώ βρίσκονται βουλευτές βουλευτές των ε, ευρωπαϊκών κρατών, ε, κράτη που πλέον ε, χαίρουν και απολάβουν αυτοδιάθεσης. Στο δικό μας το Κοινοβούλιο συνυπάρχουν διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές φυλές, διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτισμών και κρατών, όλοι όμως ενωμένοι με μία και μόνο βούληση. Η βούληση να μην επαναληφθούν στην Ήπειρό μας αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν κατά το παρελθόν. Είναι θαύμα το ότι μπορέσαμε στην Ήπειρό μας να επιτύχουμε τη συμπηλίωση μετά από όλα αυτά που έλαβαν χώρα. Για μένα λοιπόν κάθε φορά ε, είναι σαν να είναι μια καινούρια φορά να βρίσκομαι σε αυτήν την ε, αίθουσα, στην Ολομέλεια και να βλέπω ότι πλέον όλοι μας, απόλυτα ελεύθεροι, δημιουργούμε μια Ευρώπη. Πώς κατορθώνουμε τελικά να ξεπεράσουμε τη φτώχεια και να ε, ακυρώσουμε ε, φραγμούς και φυσικά εμπόδια. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε πάρα πολλά προβλήματα και σήμερα να συμβιώνουμε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Το θαύμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης σίγουρα και μπορεί να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει στο να μην επαληφθεί μια τέτοια ανθρώπινη καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως και δεν έχουμε εγγυήσει για κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορέσαμε διαμαγείας να εξολοθρεύσουμε και να ξαντραποδίσουμε τον πόλεμο από τον κόσμο. Ο πόλεμος εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν όμως πλέον οι δομές εκείνες οι οποίες παρεμποδίζουν την επαναφορά του πολέμου. Και αυτό διότι έχουμε υπερεθνικές δομές. Οποτεδήποτε και αν κατορθώνουμε να τις ε, καταστρέφουμε τις δομές αυτές, παρόλα αυτά ελοχεύει ο κίνδυνος να επανέρχεται ο εθνικισμός, ε, η διακριτική μεταχείριση, το μίσος. Μπορέσαμε βέβαια να φτιάξουμε ένα σύστημα που να παρεμποδίζει τον πόλεμο, δεν μπορέσαμε όμως να εξαφανίσουμε πλήρως τον πόλεμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη που φοβούνται τον πόλεμο, διότι δυστυχώς και πάλι μονόπλευρα μετατίθενται σύνορα στην Ήπειρό μας. Οφείλουμε λοιπόν να επαγρυπνούμε. Κυρίε και κύριοι, η ελευθερία και η ειρήνη είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της δικής μου της μεταπολεμικής γενιάς. Εγώ ως Γερμανός ανήκω σε εκείνους οι οποίοι δεν φέρουν την ε, ε, ατομική υπετιότητα γιατί γεννήθηκα μετά τον πόλεμο υπάρχει όμως μια συλλογική υπετιότητα την οποία δεν ξεχνώ όπως και όλοι εκείνοι που γνωρίζουν ότι η ειρήνη, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός Όλα αυτά μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εφόσον δεν παραμένουν κενά λόγια και μόνο εφόσον εφαρμόζονται στην πράξη. Η μεγάλη δύναμη αυτού του Κοινοβουλίου είναι ότι πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε και γι' αυτό το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη ευθύνη να αναγνωρίσει ότι η ειρήνη, η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη κάθε μέρα πρέπει να είναι αντικείμενα ε, προσπαθειών ε, και υπεράσπισης εκ μέρους μας. Γι' αυτό λοιπόν η κοινοβουλευτική συνέλευση, η δική μας, είναι ένα καλό, δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην Ευρώπη του σεβασμού και της ειρήνης. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας. Καθήκον μας λοιπόν να διαφυλάσσουμε την ειρήνη, την ε, ανεκτικότητα στην Ευρώπη και αυτό οφείλει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να προσέξετε το εξής. Επανερχόμεθα στην καθημερινότητα των εργασιών μας που σήμερα ξεκινάει με κάποιες τεχνικής φύσεως οδηγίες Σήμερα ε, έχουμε και πάλι ε, λήψη φωτογραφίες 360 μοιρών στην Ολομέλεια. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής τους συναδέλφους. Η φωτογραφία αυτή γίνεται βέβαια τμήματικά, γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλούμε την ώρα που η κάμερα είναι στραμμένη προς εσάς να στρέφετε το βλέμμα στην κάμερα και ή δυνατόν να χαμογελάτε κιόλας γιατί οι, οι φωτογραφίες αυτές θα δημοσιευθούν. Θα λοιπόν να σας ε, παρακαλέσω να παρακολουθείτε το βοηθό του φωτογράφου, ο οποίος θα σας ενημερώνει πότε η κάμερα είναι στραμμένη προς εσάς. Ε, λοιπόν, πού είναι ο βοηθός του φωτογράφου, ε, είναι ο κύριος με το άσπρο πουλόβερ. το μπέζ αυτό ο οποίος θα σας ε, κουνήσει το χέρι και θα πρέπει να ξέρετε ότι τότε πρέπει να χαμογελάσετε. Η κάμερα αυτή θα παραμείνει στην ατσία τη μέχρι την ολοκλήρωση της ε, ψηφοφορίας. Και σας παρακαλώ πολύ ε, λέει τεχνική οδηγία να μην αγγίζετε την κάμερα όταν φεύγετε. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω την οδηγία, δεν ξέρω γιατί ένα βουλευτή θα άγγιζε την κάμερα, τέλο πάντων σα το είπα. Οι φωτογραφίε λοιπόν αυτέ θα αναφερθούν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να μπουν και σε άλλε ιστοσελίδε. Που σημαίνει ότι η φωτογραφία που θα ληφθεί εδώ μπορείτε αυτή να τη χρησιμοποιείτε κι εσεί για δικού σα επικοινωνιακού σκοπού. Ελπίζω τώρα αυτέ οι τεχνικέ οδηγίε να είναι σαφεί όταν ο κύριο εδώ που σα είπα με τον Μπέζ ε, σα κουνεί στο χέρι.